Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμά σας είναι λίγο αισιόδοξο διότι οι προθεσμίες για τη μετάφραση που είναι υποχρεωτικές διότι έχουν το δικαίωμα και για τις τροπολογίες να έχουν μετάφραση οι βουλευτές δεν είναι επαρκής. Η γραμματεία μου λέει ότι η διορία κατάθεσης τροπολογιών είναι 13η Νοεμβρίου. Αυτό δεν μας επιτρέπει να ψηφίσουμε ήδη στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Αλλά θα ήθελα, αν συμπεριλαμβάνεται η έκθεση, αν δεν συμπεριλαμβάνεται μάλλον, στον κατάλογο που θα εξετάσουμε στους συντονιστές το απόγευμα για την εφαρμογή της Συνδίκης Λισαβόνας ή μάλλον αν είναι στον κατάλογο να δούμε αν είναι ρεαλιστικό και το χρονοδιάγραμμα γιατί το δίκτυο δεν έχει δουλέψει και πολύ καλά για πολλά χρόνια γιατί το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι κάτι καινούριο και υπάρχει λοιπόν σοβαρός λόγος να τα επανεξετάσουμε όλα αυτά και να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να τα χειριστεί με βάση τις διαδικασίες της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν νομίζω ότι θα υποφεληθούν οι εγκληματίε απλώς και μόνο από αυτή την καθυστέρηση. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε αν γίνεται το θέμα αυτό να λήξει μέσα στο μήνα. Αν δεν γίνεται, τότε θα αφανεί μόνο του. Αν γίνεται βέβαια ως ομάδα εμείς θέλουμε να λήξει το θέμα αν και καταλαβαίνω και της, την ανάλυση της εισηγητρίας. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές. Εδώ πρόκειται για πρόγραμμα για δίκτυο αντιμετώπισης του εγκλήματος πανευρωπαϊκά και επομένω δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα με μία και μόνη πρωτοβουλία και να ελπίζουμε ότι έτσι θα έχουμε και αποτέλεσμα. Να μην ξεχνάμε ότι μόλις τεθεί η συνθήκη ενισχύει, ακριβώς θα είναι ένα από τα θέματα όπου θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη δικαιοδοσία. Παρά λοιπόν αυτά που είπε η συγκήτρια που είναι λογικά, πρέπει να φροντίσουμε να μην τα βάλουμε όλα στο ίδιο αυτό τσουβάλι θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες να πραγματοποιηθούν αυτά που θέλει η συγγήτρια. Καταλήγω λοιπόν. Η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι αν είναι ρεαλιστικό να λήξει το θέμα πριν τη Λισαβόνα. Αν όχι, αν δεν είναι ρεαλιστικό, τότε θα ακολουθήσουμε την κανονική διαδικασία. Αν όμως είναι δυνατόν, τότε εμεί ως ομάδα συμφωνούμε να καταλήξει. και για να δείξουμε και πνεύμα, επιδείξουμε πνεύμα συνεργασίας με την Προεδρία. Δεν είμαστε κατά του να λήξει πριν τελειώσει η Προεδρία, αν και εφόσον σεβαστούν και εκείνοι τη δική μας γνωμοδότηση, το δικαίωμά μας να εκφραστούμε. Μάλιστα. Στις αρχές νομίζω θα παραμείνουμε γιατί ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και με άλλες εκθέσεις και θα τα δούμε στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών για να δούμε τι θα κάνουμε ακριβώς. Φυσικά ολόψυχα εγκρίνω αυτά που είπατε. Πράγματι είχαμε συμφωνήσει ότι πρέπει όποτε γίνεται να διεκπεραιώνονται τα θέματα γρήγορα. Μάλιστα. Πάει λοιπόν το πρώτο σημερινό θέμα. Το δεύτερο είναι η δημιουργία συνδέσμων για θέματα μετανάστευσης. Ο Ντίας Δεμίρα είναι εισηγητής, έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 30 Σεπτεμβρίου. Από τότε ο εισηγητής κυκλοφόρησε στα μέλη, μοίρασε στα μέλη ένα πρώτο σχέδιο έκθεσης και λίγη αύριο το μεσημέρι διορία κατάθεσης τροπολογιών. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ λίγος χρόνος, αλλά είχατε προειδοποιηθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση. Και στο ίδιο αυτό πνεύμα λοιπόν της ταχείας διεκπαιρέωσης και συνεργασίας, νομίζω ότι θα προλάβουν όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις τροπολογίες μέχρι αύριο το μεσημέρι. Και τώρα ο κύριος Δίας Δεμήρα και μετά η Κομισιόν και το Συμβούλιο και ύστερα οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς έχουμε μία πρόταση για τροποποίηση του 337 κανονισμού του 2004 που τροποποιεί την αρχική πρόταση για τη δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης της μετανάστευσης. Πρόκειται για μια πρακτική πολύ απλή. Θα σας αναφέρω σε λίγο όμως ποια είναι τα πιο, το, ποιο είναι το πιο ουσιαστικό περιεχόμενο. Το δίκτυο υπαλλήλων, είπαμε, δημιουργήθηκε βάσει του 337-2004 και προβλέπεται ότι οι εκπρόσωποι αυτού του οργανισμού ε, είναι αποσπασμένοι υπάλληλοι του κράτους μέλους ε, από την υπηρεσία, αποσπασμένοι υπάλληλοι της υπηρεσίας αλλοδαπών του κράτους μέλους και έχουν επαφές με τις, ε, με τους αρμόδιους οργαν... τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας υποδοχής για να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση, να βοηθήσουν στον επαναπατρισμό των ε, παρανόμων μεταναστών και να ευνοήσουν την νόμιμη μετανάστευση. Οχτώ μήνες μετά δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της λειτουργικής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, το Frontex δηλαδή. Και αυτό για να διαχειριστούμε τα εξωτερικά σύνορα και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην κατάρτιση των ε, ε, φυλάκων των συνόρων να βοηθήσουν λοιπόν στην έρευνα και στην, ε, και στην φύλαξη των εξωτερικών συνόρων λειτουργική λοιπόν συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα και να χορήγηση στα κράτη-μέλη υποδομής για την ε, κοινή οργάνωση επιχειρήσεων επαναπατρισμού. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ ζήτησα πολλές φορές να με ενημερώσουν σχετικά με τις λεπτομέρειες αυτών των κοινών επιχειρήσεων στα πλαίσια του Frontex. Λέω λοιπόν ότι έχουμε 27 κράτη-μέλη στην Ένωση και 27 αξιωματικούς συνδέσμους, υπαλλήλους συνδέσμους. Όμως στην ουσία τέτοιοι σύνδεσμοι υπάρχουν σε 133 σε 133 χώρες. Βέβαια, όλα αυτά στα πλαίσια του Frontex θα μπορούσαν να γίνουν πιο αποτελεσματικά αν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ε, μέσα στα πλαίσια του Frontex αυτούς τους αξιωματικούς συνδέσμους διότι στο Frontex δεν έχουμε καμία αντιπροσωπεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, λάβετε υπόψη σας λοιπόν αυτούς τους 133 που έχουμε ανά τον κόσμο. Η τροποποίηση του 337 θέλει ακριβώς να εκμεταλλευτούμε αυτήν την κεκτημένη εμπειρία των αξιωματικών συνδέσμων ε, στα πλαίσια του Frontex. Αυτό δεν υπήρχε στον αρχικό κανονισμό που θέλουμε να αλλάξουμε. Και η πρόταση τροποποίησης λέει ότι θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτών ε, των αξιωματικών συνδέσμων, των, υπαλλήλων, των αποσπασμένων υπαλλήλων και οι πληροφορίες να μπουν και στο δίκτυο e-Connect. Το e-Connect δεν επιτρέπει την χρήση προσωπικών δεδομένων. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τίποτα από τα προσωπικά δεδομένα. Θα μου πείτε τότε. Ε, τότε τι μας λένε όλοι αυτοί πάλι οι σύνδεσμοι, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι. Μα αναφέρονται σε μεταναστευτικές ροές, από τη χώρα υποδοχής ε, ή από διαμετακομιστικούς χώρους. Ε, ε, αναφέρεται στο μόντους operandi, στον τρόπο λειτουργίας της μαφίας, στους νέους δρόμους, στις έσοδους μετανάστευσης, αναφέρεται σε δυστυχήματα, αναφέρεται σε παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τα δίκτυα παράνομης μετανάστευσης. Ε, σε συστήματα πλαστογράφησης ε, ε, επισήμων εγγράφων. Αυτή είναι ουσιαστικά η πληροφόρηση του e σε καμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα. Εμείς επίσης θέλουμε να έχουμε πρόσβαση και στα κονδύλια του τα σχετικά κονδύλια για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, ώστε να βοηθήσουμε να ενισχύσουμε τη λειτουργία αυτού του δικτύου. Και θέλουμε να έχουμε και αυτά την παρουσίαση, να ακούμε την εξαμηνία την παρουσίαση. Και αυτά βάσει του 6.3 και του άρθρου 66 της ε, Συνθήκης ε, της ε, Ένωσης. Προτείνω λοιπόν τώρα να γίνει η εξής αλλαγή. Λοιπόν, στο 3.1 θα θέλαμε αντί να έχουμε τον όρο migration να πούμε immigration, δηλαδή μετανάστευση και όχι μεταναστευτική ροά, ροή, migration. Και μετά θέλουμε την τροποποίηση σχετικά με την ε, σύνδεση του δικτύου με το Frontex. Όπως είπε και η Πρόεδρος, δεν λέμε να γίνουν οι τροπολογίες, οι τροποποίησεις αυτές να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς εγκρίναμε ε, στις 22 Σεπτεμβρίου το μέτρο και η προθεσμία είναι 7 μέρες. 16 Νοεμβρίου λοιπόν να γίνει ψηφοφορία η πρώτη και η δεύτερη Σεπτεμβρίου, ε, Δεκεμβρίου και να περάσει από την Ολομέλεια 14 Δεκεμβρίου. Αυτά, τίποτα άλλο. Thank you very much. Um, I would like to, well, maybe first invite the, the council. Ευχαριστώ. Τώρα το Συμβούλιο, η Σουηδική Προεδρία δηλαδή. Είναι η κυρία Πέρσον, όχι. Όχι. Δεν πια είναι τότε. Τέλος πάντων η Σουηδική Προεδρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Άννα Γκέρπερ. Είμαι σύμβουλος της Προεδρίας και την εκπροσωπώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και την εισηγήτρια. Εμείς από την Προεδρία δεχόμαστε την έκθεση του κύριου Ντεμέρας γιατί συμφωνεί αρκετά με τις συζητήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο και σε προηγούμενες περιπτώσεις το Σεπτέμβριο όπου είχε συζητηθεί το θέμα η πρόταση αυτή δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες στο Συμβούλιο και καταλήξαμε ότι δεν χρειάζονται πολλές ή τεράστιες τροπολογίες. Επαναλαμβάνω ότι και οι ίδιε οι τροπολογίε του κυρίου Ντεμέρα συμφωνούν με τις προτάσεις που είχαν συζητηθεί για αλλαγές στο Συμβούλιο. Α, ευχαριστώ πολύ. Περιεκτικά μας τα είπατε. Τώρα είναι ο κύριος Ντόμπο από την Κομισιόν. Ναι, έτσι λέγομαι κυρία Πρόεδρε, τι να κάνω. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής σας για την συζήτηση αυτή, διότι εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την έκθεση και ελπίζουμε να μπορέσετε να την εγκρίνετε όσο το δυνατόν συντομότερα. Σας κατευχαριστώ, όλοι έτσι πρέπει να μιλάνε, τόσο γρήγορα, λοιπόν, τόσο σύντομα μάλλον. Ποιος έχει ζητήσει το λόγο, κύριος Κίρκοπ, ο οποίος έχει και το λόγο πρώτος. Μπορεί να σας φανεί μονότονο αυτό, αλλά και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Θα προσθέσω όμως και κάνα δυο θεματάκια. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την αίτηση, το αίτημα αυτό δημιουργίας συνδέσμων υπεύθυνων για τη μετανάστευση ιδίως στα εξωτερικά σύνορα. Ξέρω ότι με Ποιες χώρες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και άλλες το θεωρούν ιδιαίτερα λεπτό θέμα και θα έπρεπε επομένω να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις όσο γίνεται. Αλλά υπάρχει η ανησυχία μας για τους πόρους που θα διατεθούν. Γιατί όπως και με όλες τις επιχειρήσεις του Frontex λείπουν οι απαραίτητοι πόροι. Θα έπρεπε λοιπόν η κατανομή τους να γίνει καταλήλως. Όχι μόνο να υπάρχει ένα σωστό σχεδιασμό της λειτουργίας των συνδέσμων αυτών, αλλά να δοθούν και οι, ε, και οι απαραίτητοι πόροι. Βέβαια η υπηρεσία αυτή λειτουργεί μέσα στην Ένωση, αλλά οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυφθούν ιδιαίτερα για θέματα παράνομης μετανάστευσης και επιστροφών στη χώρα προέλευσης καθώς και παρανόμου εμπορίου είναι θέματα που δεν είναι μόνο εσωτερικά και γι' αυτό νομίζω ότι δεν έχουν γίνει όσα θα έπρεπε να γίνουν για να προσεγγίσουμε και κυβερνήσεις εκτός Ένωσης. Εμείς βέβαια θα αναγκαζόμαστε ούτως ή άλλως να υφιστάμεθα τις επιπτώσεις των πράξεων και ορισμένων εκτός Ένωσης. Πάντως σας συγχαίρω γενικά και θα έπρεπε να ε, τονίσω με το θέμα που ανέφερε. Ευχαριστούμε ο κύριος Ζούλτσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω τον εισηγητή Ντίας Δεμέρα διότι τα ανέλησε όπως έπρεπε τα πράγματα. Η νέα διατύπωση, μετανάστευση ή μεταναστευτική ροή, δείχνει ότι αλλάζουν τα πράγματα στην Ευρώπη στο σύνολό της, της Ένωσης. Είναι σημαντική η αλλαγή διότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται, υπονοείται η ανάγκη να αλλάξουμε και την αντιμετώπιση μας η μετανάστευση και ο εκπατρισμός θα παραμείνουν νομίζω όπως φρονώ ταπεινά χωρίς να είμαι ειδικό, κάτι το πολύπλοκο, αμφιλεγόμενο, δυναμικό και ίσως και πολύ κειμενόμενο διότι δεν θα μπορούμε να το μετρούμε σε όλες του τις διαστάσεις πάντοτε. Και άρα δεν θα είναι εύκολη η διαχείριση και αντιμετώπιση. Οι προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού που έκανε ο εισηγητής είναι τελείως απαραίτητες λοιπόν. Αναρωτιέμαι <clears throat> μήπως οι τροπολογίες θα βελτιώσουν τα πράγματα ή όχι. Παραδείγματο χάρη η καινούργια αυτή ιδέα ενός πιλωτικού ή πειραματικού προγράμματος για τον καθορισμό για την ίδρυση γραφείων του Frontex εκτός Ένωσης. Ξέρω ότι δεν θα χρειαστεί το ίδιο νομικό υπόβαθρο για αυτήν την τροπολογία όπως για την εφαρμογή γραφείων Frontex μέσα στην Ένωση. Αλλά Είναι καλή ιδέα γιατί σε χώρες όπως η Κροατία, το Μαυροβούνιο, ίσως ακόμη και η Σερβία, θα ήταν σημαντικό να υπάρξουν τέτοια γραφεία εκεί επιτόπου και σε άλλες υποψήφιες χώρες. Να συνδυαστούν δηλαδή οι λειτουργίες του Frontex και αυτών των συνδέσμων που ζητάμε. Μετά λέει ο κύριο Δία Δεμέρα, οι εξαμηνιαίε εκθέσει πρέπει να είναι πιο ελαστικές, λέει, πιο ευέλικτε. Μήπω θα μπορούσαν να είναι τριμηνιαίε αντί διότι αν είναι μικρότερη η περίοδος που θα καλύπτουν, τότε σίγουρα θα είναι πιο ευέλικτες. Αυτό είναι διαφορετικό από την αρχική πρόταση νομίζω η κυρία Κιγιόμ Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Δεμέρε. Είπατε ότι είχε γίνει μία πρώτη ανταλλαγή τον Σεπτέμβριο, ότι ήταν μία απλή έκθεση. Όμως βέβαια δεν είναι τόσο απλό γιατί υπάρχουν ερωτήσεις που θα πρέπει να διευκρινίσουμε και να απαντήσουμε. Προτείνω λοιπόν να γίνουν ορισμένες τροποποίησεις σε ορισμένα άρθρα και θα σας αναφέρω εδώ τους άξονες για τους οποίους θέλω να κάνω προτάσεις, όχι βέβαια αύριο. Είναι θέμα ορολογίας. Στην Ισπανία φάνηκε πρόσφατα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με τη μετάφραση κειμένων. Ο όρος «immigration illegal» χρησιμοποιείται πολλές φορές στο κείμενο «παράνομη μετανάστευση». Εγώ πιστεύω ότι ο όρος «migration irrégulière» ε, θα ήταν ο καλύτερος. Επίσης το, ε, το θέμα των αξιωματικών ε, συνδέσμων ε, καλύπτει και την νόμιμη μετανάστευση, όχι μόνο την μη νόμιμη. Ένας τρίτος άξονας σκέψης, ο υπάρχον κανονισμός θα πρέπει να αναφέρει και τις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους διεθνείς κανόνες για την προστασία των ετούντων άσυλο και την προστασία από το παράνομο δίκτυο διακίνησης μετανασ... παρανούς μετανάστευσης. Επίσης, ότι αυτοί οι αξιωματικοί θα πρέπει να καλούνται στις σχετικές συνεδριάσεις του Frontex και θα πρέπει επίσης να είναι υπόλογοι με μία εξάμεινη έκθεση. Εμείς ε, μιλάμε πάρα πολύ για το Frontex ε, και για τις διάφορες αποστολές, ας πούμε οργάνωση ε, των διαφόρων charter επαναπατρισμού καταναγκαστικού επαναπατρισμού. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς σε όλη αυτή την ιστορία τι είναι αυτό το οποίο διακρίνει τους αξιωματικούς ε, συνδέσμους από τους υπαλλήλους του Frontex, ο κύριος Ταβάρες. Εγώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Μία γενική και μία πιο περιθωριακή. Εγώ εδώ δεν θέλω να ξαναρχίσουμε εδώ την ιδεολογική συζήτηση αν η μετανάστευση είναι παράνομη ή άτακτη. Αλλά ε, εδώ η εισηγητής αναζήτησε να υπάρχει μία συνεκτικότητα στο κείμενο όπου μιλούσαμε για παράνομη μετανάστευση. Εμείς θα πρέπει να εγγυθούμε ορισμένους όρους που θα επιτρέπουν να καλύπτουμε όλες τις νομικές περιπτώσεις στα κράτη-μέλη Ας πούμε σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν μιλάμε για παράνομη μετανάστευση. Μην ξεκινήσουμε λοιπόν και πάλι την ιδεολογική συζήτηση αλλά από γλωσσικής πλευράς ο όρος άτακτη μετανάστευση είναι καλύτερος. Τώρα, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι θα ήταν καλό να συνεργάζονται όχι μόνο με το Frontex αλλά και με άλλα θεσμικά όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, εδώ συζητάμε εμείς για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού ασύλου. Και σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για συνεργασία αυτών των συνδέσμων με αυτόν τον οργανισμό, γιατί όλα αυτά είναι τα βασικά πιόνια του στη, στο, στη διαδικασία της μετανάστευσης. Στα κράτη-μέλη, για χρόνια αφέθηκε η μετανάστευση στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εστερικών. Και τώρα διαπίστωσαν ότι θα πρέπει να ασχοληθούν με την μετανάστευση και τα Υπουργεία εργασία, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων ή το Υπουργείο Οικονομίας κλπ. Αυτούς λοιπόν τους αξιωματικούς συνδέσμους να τους έχουμε μόνο σε συνεργασία με το Frontex χωρίς να προβλέπουμε ότι θα πρέπει ευρύτερα να αρχίσουν να συνεργάζονται και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την μετανάστευση. Νομίζω ότι δεν καλύπτει τις προσδοκίες μας. Πάντως, στο μεταξύ, συγχαίρω τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω τον εισηγητό να μας παρουσιάσει συμπεράσματά του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους όσους επένεσαν την έκθεσή μου και την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την Ανίτα Έγκμπεργκ, λέει ο, ο Λοιπόν, υπήρξε τεράστια συνένεση γύρω από αυτό το θέμα και οι 27 κράτη συμφώνησαν. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ την εκπρόσωπο του Συμβουλίου όπως και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Τώρα για την τοποθέτηση του Τίμωθη, δηλαδή του κυρίου Κίρκχοπ, πάντα εύστοχη δεδομένου ότι ήταν και υπουργό Εσωτερικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρει πολύ καλά γιατί μιλάμε. Τώρα για τα κονδύλια. Εμείς, Τίμωθη, έχουμε πολλές ελπίδες. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Το 2005 το Frontex είχε 5 εκατομμύρια ευρώ και το 2010 το Frontex και αυτό χάρη δηλαδή με τις ε, αλληλέγγυες ε, τροπολογίες σοσιαλιστών και λαϊκών ε, για τον προϋπολογισμό το Frontex ξεπερνάει τα 80 και εκατομμύρια. λοιπόν, το Frontex θα πρέπει να έχει επαρκείς ικανότητες για τη διαχείριση αυτών των νέων κονδυλίων που διαθέτουμε. Επίσης, να απαντήσω και σε άλλους συναδέλφους. Η κυρία Γκυλέμ λέει ότι θα προτείνει τις τροπολογίες της, τις οποίες εκτιμώ ιδιαίτερα και θα τις εστιάσει γύρω από τέσσερα βασικά ζητήματα και όταν μιλάει για ορολογία, να απαντάω έτσι και στον κύριο Ταβάρες που μιλάει επίσης για ορολογία. Κοιτάστε, πραγματικά, δεν θα έχετε προβλήματα με μένα γιατί εγώ είμαι υπέρμαχος της ακριβούς χρήσης της άτακτης ή λαφρέας και όχι παράνομης. Διότι εγώ θέλω να αποστηρώσω τον όρο, να μην έχει ιδεολογική χρειά. Και για Ορισμένα κράτη-μέλη, η άτακτη μετανάστευση, η λαθρομετανάστευση έχει μόνο διοικητική διάσταση και όχι ποινική, ενώ για άλλους έχει ποινική. Τώρα το κείμενο που αφορά στο Frontex και αυτό το οποίο τροποποιούμε τώρα μιλούν για παράνομη μετανάστευση. Αν αυτό λοιπόν το illegal, το παράνομο, το βάλουμε λαθρέα ή άτακτη, Εγώ δεν θα διστάσω ούτε στιγμή να δεχθώ αυτούς τους όρους. Τώρα για την εντολή αυτών των αξιωματικών συνδέσμων. Όλες αυτές οι απόλυτα λογικές διεκδικήσεις θα δημιουργήσουν πρόβλημα με τον ρόλο βάσει του 337 που έχουν αυτοί οι αξιωματικοί σύνδεσμοι. Λοιπόν, οι αρμοδιότητες τους ποιες είναι, είναι να... Είναι πρόληψη και καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Αυτοί λένε παράνομη μετανάστευση. Μετά, επαναπατρισμός των λαθρομανεσ... λαθρομεταναστών. Και τρίτον, διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης. Για να τους δώσουμε τώρα εμείς άλλες αρμοδιότητες θα πρέπει να προτείνουμε μια άλλη αλλαγή του 337. Αλλά αυτό συνηθίζεται, γιατί εμείς δεν πρέπει να είμαστε στατικοί μπροστά σε ένα νομοθετικό κείμενο. Πρέπει να το μεταρρυθμίζουμε κάθε φορά που μπορούμε. Ο κύριος Σταβάρης και η κυρία Γκυλέμ μίλησαν για το άσυλο. Και το άσυλο είναι ένα θέμα γύρω από το οποίο δεσμευόμαστε ιδιαίτερα. Εμείς παραπονεθήκαμε για την ε, αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά τη γνώμη μας, ότι δηλαδή για το ότι θα έπρεπε το 2010 να έχουμε μια κοινή πολιτική ασύλου. Και εμείς είπαμε, μάλλον και εκφράσαμε την λύπη μας ότι από το Ταμείο Προσφύγων πήραν λεφτά για να δημιουργήσουν τον οργανισμό για το ευρωπαϊκό άσυλο. Όμως το δίκτυο των αξιωματικών συνδέσμων όπως ανέφερα προηγουμένως δεν έχει αρμοδιότητες για θέματα ασύλου. Λοιπόν. Και όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι αυτονόητο, είναι απαραίτητο να προασπίσουμε το πρωτογενές δίκαιο. Εγώ τις τροπολογίες θα τις εξετάσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα προσπαθήσω να έχω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση γύρω από την έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, μου λένε ότι προβλέπεται για την πρώτη ψηφοφορία στην Επιτροπή και μέσα Δεκεμβρίου για την Ολομέλεια. Αλλά κοιτώντα το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσαμε να έχουμε λίγε περισσότερε μέρε ε, για να μπορούν να υποβληθούν ε, ε, οι τροπολογίε. Συμφωνείτε την επόμενη Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Ναι, εμένα μου φαίνεται εντάξει την ε, Τρίτη, αλλιώς ε, αν δεν γίνεται την επόμενη Τρίτη. Εγώ θέλω να γίνει συζήτηση και μπορώ να αφήσω ανοιχτή την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ωραία, οπότε ορίζουμε την ε, προθεσμία για τις 10 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, σε 15 λεπτά προβλέπεται η ψηφοφορία, συνάδελφοι, σύμφωνα με την μοιρασία διάταξη. Θέλω να πάω να διακόψουμε τη συνεδρία συνεδρίαση 15 λεπτά για να μπορείτε να περάσετε στα γραφεία σας αν χρειάζεται και να πάρετε τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική πλησιοφορία. Ο κύριος μας είπε έχει όμως κάτι διαδικαστικό να μας παρουσιάσει. Πρόεδρε, μια που έχουμε χρόνο, θα ήθελα να πω όσοι είμαστε μέλη της Επιτροπής για τις ε, πτήσεις ε, της CIA Είμαστε ιδιαίτερα ενοχλημένοι από αυτές τις δίκες, ε, ε, τις αποφάσεις μάλλον στην Ιταλία. Για τις δύο καταδίκες λοιπόν στην Ιταλία και θέλω να θυμηθώ εδώ και τον Κλάουδιο Φάβα που ήταν τότε πρόεδρος ε, και τον συνάδελφο Κάρλο Κοέλιο. Είναι πολύ θετικά αυτά τα νέα. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, διακόπτουμε τώρα. Δέκα και μισή θα επανέλθουμε με τις κάρτες ψηφοφορίας παρακαλώ.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

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Colleagues, can I ask you all to sit down so we can start the vote? Can, can, colleagues, can we please sit down and we can start the vote and our conversation? Παρακαλώ να ψηφίσουμε αν έχετε ιδιωτικές συνομιλίες να τις κάνετε απ' έξω. Άψογα κάθισαν όλοι. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες. Η δική μου πάντως δεν δουλεύει. Αν είστε όλοι έτοιμοι και όλες, ξέρω ότι κάποιος δεν την έχει αλλά την φέρνουνε μου είπανε. Μάλιστα. Έτοιμοι. Μία μόνο ψηφοφορία για μία έκθεση γιατί οι άλλοι έχει βγει από την ημερήσια διάταξη. Θα ψηφίσουμε λοιπόν για την έκθεση του Αλεξάνδρου Αλβάρο. Ορίστε κύριε Ντεμίρα. Ένα διαδικαστικό κύριε μου. Αυτό το σύρμα με ανησυχεί ιδιαίτερα. Διότι αυτό σημαίνει ότι το, η συσκευή ψηφοφορίας δεν είναι συνδεδεμένη. Λάβετε το υπόψη σας. κατανοώ. Εγώ όμως είμαι πολύ κακή με τις νέες τεχνολογίες. Δεν αλλάζετε θέση καλύτερα. Κοιτάξτε, το πρωί όταν μπήκα ήταν μια ομάδα που μου είπε «Καλημέρα σας κυρία, είναι είμαστε της Αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας». Τι να σημαίνει άραγε αυτό, έχει καμία σχέση με το ευγάλσιμο των σειρμάτων. Α, και άλλο διαδικαστικό, κύριος Μπουσουτσίλ. Ναι, συντομότατα. Φαίνεται ότι λόγω των αλλαγών της ημερήσιας διάταξης εχθές έχουν συγχυστεί μερικοί συνάδελφοι και νόμιζαν ότι η συνάντησή μας άρχιζε τώρα ενώ έχουμε δουλέψει ως κανονική συνεδρίαση για εδώ μια και μια μισή ώρα. Ίσως στο μέλλον να ανακοινώνονται οι αλλαγές σαφέστερα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γιατί οι περισσότεροι δεν ήρθαν για αυτόν τον λόγο. Συμφωνώ απόλυτα και το σημειώνω θα το στείλω στη γραμματεία και τον πρόεδρο. Εγώ το είπα χθε βέβαια σε όποιον ήταν παρόν, αλλά δεν ήταν όλοι και όσοι δεν ήταν παρόντες πρέπει να έχουν και αυτοί έναν τρόπο να μαθαίνουν τις αλλαγές, σύμφωνοι. Λοιπόν, έτοιμοι για την ψηφοφορία. Παρακαλώ να έχετε υπομονή γιατί είναι η πρώτη φορά που διευθύνω ψηφοφορία. Λοιπόν, έκθεση Αλεξάνδρου Αλβάρο για γαλλική πρωτοβουλία για να εγκριθεί με του Συμβουλίου για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνιακό τομέα. Πρώτα, μια η τροπολογία 85 για απόρριψη συνολική της πρότασης. Αν εγκριθεί αυτή καταπίπτουν όλες. Όποιοι ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας αυτής. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τις υπόλοιπες. 7 υπέρ. κατά Χες. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. κατά Χες. Από Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. 10 υπέρ Κατά. ποιες εγκρίνεται 11 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 12 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται τροπολογία 91 υπέρ κατά ποιες Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Α, έλεγχος ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 91 προς το σημείο 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι και όλες. Λίγοι. 26 υπέρ 14 ε, κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται όντως. Δεν βλέπει. Α, καλά, θα το σημειώσουμε. Ότι ψηφίσατε υπέρ. 27 υπέρ. 92 λοιπόν. υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Όχι 13, 93 της λέει η γραμματεία. Α, 93 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται 13 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται και τώρα η 94 με προφορική τροποποίηση με την τροποποίηση υπέρ κάποια σύγχυση όχι Α, ωραία. υπέρ λοιπόν κατά ποιες απορρίπτεται 17 υπέρ κατά yes. εγκρίνεται 95 υπέρ τα yes. απορρίπτεται 96 υπέρ κατά yes. εγκρίνεται 97 υπέρ κατά υπέρ απορρίπτεται 98 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 18 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 99 υπέρ κατά χοχές επαλήθευση τροπολογία 99 προς το σημείο επετά ψήφισαν όλοι και όλες μάλιστα τότε λίγη ψηφοφορία υπέρ 28 κατά 15 εγκρίνεται η 19 έχει αποσυρθεί 20 κατά τμήματα πρώτο τμήμα, ο, εκείνο δηλαδή χωρίς την έκφραση Europol και Eurojust, υπέρ. Τα, yes. εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα δηλαδή Europol και Eurojust υπέρ, κατά, yes. εγκρίνεται και αυτό. 100 υπέρ, τα, επαλήθευση. Τροπολογία 100, 15 υπέρ 9 κατά. όχι, τώρα αρχίζει η τροπολογία για την 100, τώρα. Μην νομίζετε, δεν τα κανονίζω εγώ όλα αυτά, λοιπόν τέλος. όλοι και όλες. Μάλιστα. 25 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται 21 υπέρ κατά yes εγκρίνεται 22 υπέρ τα yes εγκρίνεται 101 υπέρ τα yes εγκρίνεται 27 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 102 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 28 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 103 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 29 υπέρ κατά χες νομίζω ότι εγκρίθηκε εγκρίνεται εγκρίνεται 30 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ α εγκρίνεται 33 υπέρ τα αποχές εγκρίνεται 34 με προφορική τροποποίηση υπέρ με την τροποποίηση υπέρ τα χες επαλήθευση 34 με την προφορική της τροποποίηση 23 υπέρ 18 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται Άρα καταπίπτει 106. 35 πάλι με προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. Αλλά ίσως να επαληθεύσουμε για να είμαστε και σίγουροι. Η 35 με προφορική τροποποίηση αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι και όλες. Λίγοι. 24 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται πράγματι 107 καταπίπτει 36 ε, και οι 108 ταυτόσημες μαζί υπέρ κατά χες εγκρίνονται 37 37 υπέρ κατά χες Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Τα. Χες. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά ποιες γκρίνεται 41 υπέρ κατά ποιες γκρίνεται 42 υπέρ κατά ποιες επαλήθευση 42 27 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται 43 υπέρ κατά χέρες εγκρίνεται 44 υπέρ κατά χέρες εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε αλλά θα επαληθεύσουμε την 47 άρχεται η ψηφοφορία ήρθαν όλοι Έληξε η ψηφοφορία. Όντως απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Τα. Τες. Απορρίπτεται και αυτή. 49. Υπέρ. Τα. Τες. Εγκρίνεται. Άρα καταπληκτή 113. 50. Πώς, πώς. Σχόλια. 50. Υπέρ. Κατά. Ποιες. Απορρίφθηκε. 51 υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Ποιες. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 117 με προφορική τροποποίηση. Υπέρ. 117 υπέρ με την προφορική τροποποίηση. Κατά. Ποιες απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά ξέρεις, εγκρίνεται 50 Για πέστε μου, νομίζετε ότι μπορούμε από την 54 μέχρι την 63 να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. 62, ναι, μέχρι την 62. 54 με 62 υπέρ κατά πάχες εγκρίνονται 63 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε καλύτερα για την 63 ηλεκτρονική ψηφοφορία Has everybody voted? Yep, vote's closed. Πέραση ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 118 υπέρ. Those against. Κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά, αποχές. Μάλλον είναι κρίθερα για να ελέγξουμε. 67. Vote is open. Everybody voted. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 18 κατά, Είναι κρίθη. 64. Τι 119 Α, καταπίπτει, ναι. 64, λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να να ελέγξουμε, αν θέλετε. Για την 64, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ, άρχιτε ψηφοφορία. 64. 64. Vote is closed. Πέρασε ναι, ναι, πραγματικά. 23 προς 21. Πολύ μικρή πλειοψηφία. Τροπολογία 68, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 69, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 70 με προφορική τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, μέχρι την 84 όλες μαζί, εντάξει. 71 έως 84 συμπεριλαμβανόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κάποια σύγχυση νομίζω υπάρχει, αλλά τώρα ψηφίσαμε. Θεολογικές σκέψεις. 3. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 καταπίπτει. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 2 και οι 3 έχουν αποσυρθεί. Οι 4 υπέρ. Οι 4 λέω υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 σε δύο τμήματα. Έχει το κείμενο μπροστά σας νομίζω, δεν θα σας το διαβάσω. Το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 88. Α, Α, επειδή είναι κρίθη η τροπολογία 5, θα ψηφίσουμε μόνο το, τη δεύτερη πρόταση του 88. Λοιπόν, αν είχε απορριφθεί η 5 θα ισχύει η καταπληκτική ψηφοφορία που δεν ισχύει. Τώρα έχουμε μόνο μία ψηφοφορία για τη δεύτερη πρόταση του 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Does Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίες. Με μεγάλη ψηφία εγκρίνεται 36 υπέρ, 2, αποχε... 2 κατά και 7 αποχές. Συγχαρητήρια στον συγητή. Okay. <laughs> My maiden vote went well. Thank you. <laughs> Η πρώτη μου ψηφοφορία πήγε πολύ καλά. Μπράβο, σας ευχαριστώ. can I, can I ask you to leave the room? Σας παρακαλώ να βγείτε με ησυχία από την αίθουσα, συνάδελφοι. Can those who want to talk... Όσοι θέλουν να μιλήσουν να το πράξουν απ' έξω. Δεν θέλω πηγαδάκια. Γιατί έχουμε και άλλη ημερήσια διάταξη. Και το επόμενο θέμα, το 11 δηλαδή, Πρέπει να σας πω πριν το εξετάσουμε ότι η Ιταλική τηλεόραση είναι παρούσα εδώ και κινηματογραφή του συναδέλφου. Α, όχι, του Κοινοβουλίου είναι λέει. Α, μάλιστα. Το 11 λοιπόν, το 11 η μεταφορά των διαδικασιών σε ποινικέ υποθέσεις. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μπένοβα. Ελπίζω να το προέφερα σωστά. Um, Μου δίνουν οδηγίε εδώ γι' αυτό αργό λοιπόν. Η συζήτηση στο Συμβούλιο για την πρόταση αυτή συνεχίζεται και δεν αναμένεται σύντομη απόφαση. Παρακαλώ ησυχία συνάδελφοι, τι κατάσταση είναι αυτή. Όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Είναι πρόταση τρίτου πυλώνα που θα επηρεαστεί πολύ όπως και άλλες βέβαια από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, δεν φαίνεται πιθανό να δημοσιευτεί στην ε, επίσημη εφημερίδα πριν από τον επόμενο μήνα και μπορεί να ξαναρχίσει η διαδικασία από την αρχή σύμφωνα με τους κανόνες της συναπόφασης. Θα συμπεριληφθεί βέβαια στον κατάλογο των διαδικασιών που θα συζητήσουμε το απόγευμα με τους συντονιστάς. Η εισηγήτρια κυρία Μόνικα Κεμπένοβα έχει το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω αυτά που είπατε. Η θέση μου ως προς την πρωτοβολία αυτή είναι γνωστή εδώ και καιρό. Νομίζω ότι είναι πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για να πετύχουμε την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην διεκπαιρέωση των εγκληματικών υποθέσεων με προάσπιση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων. Έχω κάνει μια εισαγωγή στην έκθεσή μου, αλλά τελικά το σχέδιο έκθεσης έχει γίνει γνωστό σε όλους σας, δυστυχώς βέβαια μόνο στα αγγλικά. Αυτό οφείλεται στην πίεση χρόνου που υποστήκαμε στη διαδικασία αυτή. Δεν έχουμε ακόμη το τελικό κείμενο του Συμβουλίου διότι την Τετάρτη μόλις έληξε η τελευταία συνεδρίαση. Μερικές χώρες, Ιταλία, Πορτογαλία, το Βέλγιο και άλλες, διαφώνησαν με τη συζήτηση στην ομάδα εργασίας, διαφώνησαν να λήξει η διαδικασία. Και γι' αυτό μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα για τη λήψη και τη τελική απόφαση καθυστερήσει δηλαδή. Και όταν θα τεθεί ενισχύει την 1η Δεκεμβρίου η συνθήκη της Λισαβόνας, η συνθηκη τη λισαβονα ολόκληρη θα καταργηθεί αυτή. Εκτός αν έχει δημοσιευθεί στην, στην επίσημη εφημερίδα μέχρι τις 31 Νοεμβρίου. Πρέπει λοιπόν να ομολογήσω ότι η κατάσταση στο σημαντικό αυτό τομέα της ε, πολιτικής καταπολέμησης του εγκλήματος δεν είναι και πολύ ενθαρρυντική. Σκεπτόμενοι λοιπόν τις αρνητικές αυτές συνέπειες που θα έχει επί της διαδικασίας η αλλαγή, θα ήθελα να προτείνω να εγκρίνει το Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα Ερωτώ λοιπόν το Συμβούλιο. Σχεδιάζουν να εγκρίνουν στη συνεδρίασή τους στις 30 Νοεμβρίου την προτινόμενη διατύπωση. Εάν όχι τότε ολόκληρη αυτή η διαδικασία για τους λόγους που σας ανέφερα δεν θα ισχύσει. Και άρα θα χρειαστεί νέα πρωτοβουλία από άλλα χώρες μέλη και την ίδια με βάση πλέον τη συνθήκη της Λισαβόνας για να μην σπαταληθεί, να μην χαθεί όλη αυτή η εργασία που έγινε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα μια σαφή θέση εκ μέρους του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπένοβα. Μου λένε ότι το Συμβούλιο απουσιάζει. Α, η Κομισιόν μόλις κατέφθασε. Θα δώσω πρώτα το λόγο σε όσους συναδέλφους τον ζήτησαν, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστότερο. Και εντωμεταξύ η Κομισιόν, ίσως και το Συμβούλιο, να μπορέσουν να ετοιμαστούν για να δώσουν κάποια απάντηση. Mm-hmm. Κυρία Βέντε. Ναι, εγώ υποστηρίζω πλήρως τη στάση της κυρίας Μπένοβα. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε ποιες είναι οι προθέσεις του Συμβουλίου. Ταυτόχρονα όμως, για να τα λέμε και ειλικρινά, η δική μας γνωμοδότηση υποτίθεται ότι θα εγκρινόταν στις 17 Δεκεμβρίου, άρα σίγουρα αφού θα έχει τεθεί ενισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Άρα τουλάχιστον για τέτοια θέματα πρέπει το Συμβούλιο να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ δεν αναμένω νέα πρωτοβουλία των χωρών μελών, αλλά από την Κομισιόν η οποία θα έπρεπε κανονικά πολλά παρόμοια θέματα όπως και για τις αντικρουόμενες νομοθεσίες κτλ. να τα θέσει επί νέας Αν όχι, αλλιώς, τότε όλη αυτή η ιδέα του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και λοιπά που είναι τόσο ωραία στα λόγια δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Εκτός αυτού, λόγω του ότι αυτές οι πρωτοβουλίες ε, αυτή η συγκεκριμένη προέρχεται από 16 χώρες μέλη σχεδόν από όλο το Συμβούλιο δηλαδή αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τους ίσως για αυτόν τον λόγο τίποτε από αυτά που τους λέμε εμείς στο Κοινοβούλιο. Και αυτό δεν είναι σωστό. Σωστός τρόπος νομοθέτησης. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι ακόμη είναι άδειε οι καρέκλες, οι πολυθρόνες του Συμβουλίου, τότε να μας το σχολιάσει η Κομισιόν, δεν ξέρω ποιος ή ποια, η κυρία Εύα Τσαμαριάν. Καλημέρα σα, κύριε Πρέμ. Ζητώ συγγνώμη που ήρθα τόσο αργά. Δυστυχώ δεν πρόφτασα να ακούσω όλη την εισαγωγή τη εισηγήτρια. Αλλά νομίζω ότι ελέγχθη ότι δεν θα πρέπει η πρόταση αυτή να περάσει τόσο βεβαιασμένα και να υπάρχει λίγος περισσότερος χρόνος. Προς το παρόν, αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει η Προεδρία γιατί ξέρω ότι η Προεδρία ενδιαφέρεται να ολοκληρώσει την πρόταση αυτή πριν από το τέλος της Προεδρίας. Δεν θα πρέπει εγώ λοιπόν να απαντήσω εδώ. Εάν δεν συμβεί αυτό πριν από το τέλη της Προεδρίας, θα υπάρχει μια νέα κατάσταση, γιατί εντωμεταξύ θα έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Και τότε η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει καινούρια πρόταση και αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο. Εάν δεν υιοθετηθεί όμως από το Συμβούλιο μέχρι τα τέλη του έτους, δεν θα υποβάλει μια πρόταση Κομισιόν. Γιατί μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε κατά πόσο θα γίνει δεκτή η πρόταση όχι. Ε, και θα πρέπει η Κομισιόν μετά να έχει κάποιο καιρό για να υποβάλει την καινούργια πρόταση. Καταλαβαίνω ότι ίσως είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα αλλά όλα αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από την Σουηδική Προεδρία. Εάν δεν ολοκληρωθεί, λέω, μέχρι τα τέλη του έτους, η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποβάλει μια καινούρια πρόταση. Αλλά θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση των επιπτώσεων και μετά να αποφασιστεί προσεκτικά ποια θα είναι η καλύτερη κατεύθυνση που θα πρέπει να αναλυφθεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ νομίζω μπορεί να εξηγηθεί η απουσία της, ε, του Συμβουλίου από το γεγονό ότι κάπως ε, έχουμε βιαστεί. Τι να σας πω. Α, ας είχαν κάποιον να μπορεί να τους ειδοποιήσει ότι έχουμε προχωρήσει. Και τώρα δεν έχουμε απάντηση. Ε, καταλαβαίνω. Χωρίς απάντηση είναι δύσκολο να πούμε θα κάνουμε εμείς. Αλλά οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο που θα συζητήσουν οι συντονιστές σήμερα το απόγευμα. Και αν κατάλαβα το, την εισηγήτρια σωστά, μάλλον δεν θα συμφωνήσει έτσι κι αλλιώ το Συμβούλιο. Ε, βέβαια, αν κοιτάξετε πόσα πράγματα πρέπει να έχουν αποφασίσει μέχρι τα τέλη Νευρίου, θα πρέπει 24 ώρες το 23 να συνεδριάζουν. Έχετε κάποια πρόταση για δικασία, κυρία τη Εγώ θα έλεγα θα πρέπει να περιμένουμε τη συνεδρίαση το απόγευμα. Και θα ήθελα να αναφέρω, ο χωρίς την τοποθέτηση του Συμβουλίου, εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τίποτα. Θα πρέπει να ακούσουμε κατά πόσον η απόφαση του Συμβουλίου θα είναι για τις 30 Νοεμβρίου ή όχι. Χωρίς να το ξέρουμε αυτό δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τίποτα ε, τότε προτείνω, γιατί φαίνεται ότι η Σουηδική Προεδρία ξυπάστηκε, ξαφνιάστηκε. Προτείνω λοιπόν μετά από τον κύριο Μπουσουτήλ να το αφήσουμε το θέμα, να περιμένουμε την απάντηση του Συμβουλίου όποτε και αν έρθει να συνεχίσουμε ίσως το απόγευμα ή το βράδυ με τους συντονιστές. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ναι, αυτό και εγώ ακριβώς θα έλεγα. Ακριβώς το Συμβούλιο να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στους συναδέλφους του, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου εδώ, έτσι ώστε να μπορούμε το απόγευμα στους συντονιστές να το συζητήσουμε. Καλό θα ήταν να το μεταβιβάσει ο εκπρόσωπος. Ωραία, η κυρία Βέμπερ. Μάλιστα. Και αν το Συμβούλιο πει ότι ναι, αλλά μέχρι το τέλος του, ναι, ναι, ναι, μέχρι το τέλος του μήνα θα τα έχουμε γκρίνει όλα, θα είναι όλα πολύ καλά. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό σημαίνει και σε αυτή την περίπτωση ότι είναι άχρηστη όλη μας η δουλειά. Διότι η έκθεση και οι τροπολογίες δεν θα ληφθούν υπόψη από το Συμβούλιο. Κατάλαβα ότι η Κομισιόν είπε ότι αν χρειαστεί να υποβάλει πρόταση θα το κάνει με την τέουσα διαδικασία, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν είναι σωστό να έχουμε μια κακή νομοθεσία, χειρότερα από το τίποτα είναι. Να περιμένουμε για να καταλήξουμε σε κάτι λογικό και συνεπές. Ό,τι και να πει λοιπόν το Συμβούλιο για το απόγευμα, Νομίζω ότι στους συντονιστές μπορούμε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, ό,τι και να πει το Συμβούλιο. Αυτό ισχύει για πολλές εκκρεμούσες διαδικασίες. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Μα ακριβώς αυτό είναι το θέμα που πρέπει να συζητήσουν οι συντονιστές. Δηλαδή, αν μπορούμε να καταλήξουμε μέσα στο μήνα, τότε συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες ότι θα ήταν καλό να γίνει αυτό. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε το απόγευμα. Ακριβώς λοιπόν. Παρακαλώ κυρία Αμπένοβα με το μικρόφωνο. Ε. Ήθελα να πω ότι αν όχι τότε πρέπει να προετοιμάσουμε κοινοβουλευτικό ψήφισμα για όλες αυτές τις εκκρεμούσες περιπτώσεις. Μάλιστα θα τα πούν αυτά οι συντονιστές για όλες τις εκκρεμούσες διαδικασίες. Λοιπόν, ωραία. Τότε τελειώσαμε έληξε, εξαντλήθηκε η μερίσια διάταξη δυστυχώς. Α, μετά την κυρία Αλφάνο θα διακόψουμε μέχρι το απόγευμα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είναι πρώτη φορά που λέει αυτό το πράγμα ο κύριος Μπουσουτήλ ότι δηλαδή όλα πρέπει να τα συζητάνε οι συντονιστές. Μα και η Επιτροπή η ίδια πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο. Εμείς δεν θα μάθουμε τίποτα. Μα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και αυτόν θα τον κάνουν οι συντονιστέ. Για να τα δούμε όλα μαζί. Είναι καλύτερα να τα συζητήσουμε λιγότεροι και μετά φυσικά θα σας τα γνωστοποιήσουμε και εσάς. Ωραία ησύχασαν όλοι και όλες. Τι συμβαίνει κύριε Κροτσέτα, είναι τίποτα επίγον. Κοιτάξτε, πολύ συχνά ακούμε την έκφραση συντονιστές εδώ μέσα. Καλό είναι να τα συζητάνε οι συντονιστές, αλλά όχι κάθε φορά που τίθεται ένα θέμα να λέμε ας, τα πούν οι συντονιστές. Αν αρχίσουμε κάποιο θέμα πρέπει να ακούσουμε και τους συναδέλφους. Εδώ έχουμε πλήρη διαφάνεια, συμμετοχικότητα, δημοκρατία, ελευθερία κτλ. Το απόγευμα θα τα πούμε. Ευχαριστώ συνάδελφοι και συνάδελφε. Sì, però non mi piace che lei dica